Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη χαρά για εμένα, είναι τιμή κυρίε και κύριοι το ότι μπορώ να σας ανακοινώσω η διάσκεψη των προέδρων, το ότι η διάσκεψη των προέδρων αποφάσισε ομοφώνα να τιμήσει την κυρία Μαλάλα Γιουζαφσάη με το βραβείο Ζαχάροφ. Κυρίε και κύριοι, η Μαλάλα είναι ένα κοριτσάκι, όλοι ξέρετε την ιστορία της. Ένα κορίτσι το οποίο ε, μεγάλωνε σε μια κοιλάδα του Πακιστάν και είχε το θάρρος σε ένα ανδροκρατούμενο και βίαιο περιβάλλον να πει εγώ θα πάω στο σχολείο θέλω να μάθω γράμματα. Είμαι ένα κορίτσι και είμαι και εγώ ισότιμο μέλος αυτής της κοινωνίας. Το παράδειγμά της. Ενθάρρυνε και άλλα κορίτσια. Μια σειρά πολλά νεαρά κορίτσια να μην φοβηθούν. Και αυτό οδήγησε στο ότι φρικτοί εγκληματίες, ανθρώπους στους οποίους πρέπει να περιφρονούμε, την πυροβόλησαν με σκοπό να δολοφονήσουν. Αλλά όχι μόνο για να δολοφονήσουν τη Μαλάλα, αλλά αυτό το οποίο εκπροσωπούσε. Δόξα του Θεό, το κοριτσάκι αυτό επέζησε. Και οποιοδήποτε παρακολούθησε την πορεία της και είδε πως αυτό το κοριτσάκι μετά την ανάρρωσή του. Συνέχισε τον αγώνα της χωρίς να φοβηθεί. Αντιθέτως ενθαρρύνθηκε να συνεχίσει αυτό τον αγώνα τους. Δεν μπορεί παρά να θαυμάσει αυτή την νεαρή κοπέλα. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αρμόδια Επιτροπή και την διάσκεψη των Προέδρων για την απόφαση αυτή. Η απόφαση να βραβεύσουμε τη Μαλάλα είναι μια απόφαση που αφορά το κορίτσι αυτό, αλλά είναι και μια απόφαση για μια στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι οπουδήποτε στον κόσμο άνδρες και γυναίκες είναι ίσοι και πως όλα τα κορίτσια στον κόσμο που παλεύουν για τα δικαιώματά τους έχουν έναν σύμμαχο στο πλευρό του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Είμαι υπερήφανος γι' αυτό, για την απόφαση αυτή και χαίρομαι, πιστεύω όλοι χαιρόμαστε και πραγματικά αναμένω με ανυπομονησία να έρθει εδώ πέρα το Νοέμβριο η κοπέλα αυτή για να της δώσουμε αυτό το βραβείο. Νομίζω θα είναι πραγματικά μια σημαντική στιγμή στην ιστορία του Κοινοβουλίου και θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Πως ο αγώνας αυτής της κοπέλας δεν είναι αγώνας που συγκρίνεται με αυτά τα οποία κάνουμε εμείς εδώ. Όχι για μια κοπελίτσα που πήγαν να τη δολοφονήσουν. Μια εντεκάχρονη που της είπανε θα σε σκοτώσουμε γιατί θέλεις να πας σχολείο. Το τι θάρρος χρειάζεται για να υψώσει το ανάστημά της. Για μένα ήδη είναι μια μεγάλη προσωπικότητα του 21ου αιώνα η Μαλάλα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα για 11 φορά έχουμε την Διεθνή ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Εδώ και δεκαετίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ της κατάργησης θανατικής ποινής σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι είναι πεπισμένοι πως όσο φρικτά και αν είναι τα εγκλήματα κάποιου δεν επιτρέπεται να υπάρξει